Uh, Ευχαριστώ συνάδελφοι. Θα σας παρακαλούσα να αποχωρήσετε για να αρχίσουν οι επεξηγήσεις ψήφου. Ευχαριστώ συνάδελφε. Λοιπόν, αρχίζω τώρα εξήγηση ψήφου. Θα δώσω το λόγο για ένα λεπτό στον κύριο Μάουλου. Είναι παρόν. Παρακαλώ. Mr. Malou. Malou, 664. I go up? Αποουσιάζει. Ο κύριος Γκουτιέρεθ Πριέτο τότε. Ευχαριστώ πρόεδρε. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζήτησε μια ισχυρή νομοθετική παρέμβαση σήμερα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να προστατεύσει τα εμπορικά σήματα και ιδιαίτερα ε, την τόπια ε, ε, παραγωγή, τη μικρή βιοτεχνική παραγωγή ε, με γεωγραφική προέλευση. Γι' αυτό χρειάζεται ε, προστασία νομοθετική για να μην εξαφανιστούν. Είναι χιλιάδες οι θέσεις εργασίας, οι πολίτες, ε, οι εργαζόμενοι που χρειάζονται αυτή τη νομοθετική δράση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να διατηρηθεί η παραγωγή σε περιοχές υπαίθρου. Αυτό το σήμα Made in έχει οδηγηθεί σε εμπλοκή στο Συμβούλιο η γεωγραφική ονομασία προστατευόμενη και για μη γεωργικά προϊόντα είναι ο μόνος τρόπος που έχουν για να προστατεύουν αυτά τα προϊόντα. Σχεδόν ομόφωνα αποφάσισε σήμερα το Κοινοβούλιο την προστασία αυτών των προϊόντων. Κάντε το αυτό στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προστατεύστε ε, τους ε, μικρομεσαίους βιοτέχνες από αθέμητο ανταγωνισμό από άλλη πλευρά του κόσμου που τους πλήττει ακριβώς εκεί που τους πονάει περισσότερο, που είναι η ποιότητα και η τοπική ε, χειροτεχνία και βιοτεχνία. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η κυρία Σοντρόβα για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα και εγώ να έξω για ποιο λόγο ψήφισα υπέρ της έκθεσης κυρίας Ροζιέρ για την δυνατή αυτή επέκταση της ε, προστασίας γεωγραφικής ονομασίας. Πιστεύω πως είναι ένα καθήκον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, και θα έπρεπε να μας παρουσιάσει μια νομοθετική πρόταση για την προστασία μη γεωργικών προϊόντων. Είναι σημαντικό, είναι χρήσιμο και απολύτως απαραίτητο έτσι ώστε η μικροβιοτεχνία, η παραδοσιακή μικροβιοτεχνία να προστατευτεί. θα πρέπει αυτή η γεωγραφική ένδειξη να στηριχθεί λαμβάνοντας υπόψη την παραδοσιακή γνώση που θα προστατεύσει και θα πρέπει αυτό να περιγραφεί επαρκώς. Για παράδειγμα, επαγγελματική κατάρτιση. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τονίζει πως έχει σημασία να επενδύσουμε εκεί και απευθύνει μια έκκληση στα κράτη-μέλη να χρησιμοποιήσουν τη δυνατότητα οικονομικής στήριξης στο θέμα αυτό. Η κυρία Στέγκλερ, ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να συγχαρώ τη Βιρζινή Ροζιέρ για το καταπληκτικό αποτέλεσμα. 608 ε, ψήφοι, δηλαδή 628 βουλευτές είναι υπέρ της επέκτασης ε, της προστασίας γεωγραφικής έδειξης και σε μη, γεωργικά προϊόντα και στη Σκωτία έχουμε κάποια τοπικά προϊόντα που θα υποφεληθούν πολύ από μια τέτοια πιθανή επέκταση γιατί στον παγκοσμιοποιημένο κόσμο έχουμε πολύ μεγαλύτερες προκλήσεις με τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ε, γι' αυτό είμαστε ευγνώμενοι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στην κυρία Ροζιέβα, για την έκθεσή τη, αλλά χαίρομαι ιδιαίτερω γιατί η συντριπτική πλειοψηφία των Ευρωβουλευτών τάχθηκε υπέρ τη επέκταση τη Προστασία γεωγραφική ε, ένδειξη και σε μη γεωργικά προϊόντα. Η πρόκληση ανήκει τώρα και τον Παλάκη βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει πρόταση. Ξέρετε ότι το Κοινοβούλιο είναι υπέρ θα δώσει κάποια συνέχεια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη-μέλη στο Συμβούλιο. Ευχαριστώ κυρία Νίνα Γκίλ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η δημιουργία ενό πανευρωπαϊκού συστήματο προστασία ε, ε, γεωγραφική ένδειξη ήδη έχει δείξει πόσο ζωτική σημασία είναι για πολλά γεωργικά προϊόντα. Τώρα είναι επίση ζωτικό να ε, επεκταθεί για να καλυφθούν και άλλα αυθεντικά προϊόντα. Είναι κατακαιρματισμένη σήμερα η κατάσταση, όπου κάποια κράτη-μέλη δεν προσφέρουν την παραμικρή προστασία, ενώ έχουν και πολύ αποκλίνοντες ορισμούς. Ε, είναι πολύ σημαντικό να προστατεύονται οι χώροι παραγωγή, τοπική παραγωγή. Γι' αυτό σήμερα υπερψήφισα την έκθεση αυτή για την επέκταση της γεωγραφικής ένταξης σε μη γεωργικά προϊόντα. Εγώ είμαι από ε, τα δυτικά Midlands και έχουμε πάρα πολύ καλά προϊόντα πορσελάνης και ε, θα πρέπει να ε, κάνουμε ό,τι μπορούμε έτσι ώστε ε, να προστατεύονται και να μην ε, ε, εξωθούνται από την αγορά από φθηνές απομιμήσεις. Χρειάζεται λοιπόν ειδική προστασία. Ευχαριστώ, η κυρία Μουρβάη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ πρέπει να σας πω ότι υποστήριξα την έκθεση αυτή. Για ποιο λόγο. Να σας εξηγήσω. Στην Ουγγαρία έχουμε κάποιους κανόνες που ισχύουν για αυτά τα προϊόντα. Ε, και η νομοθεσία στην Ουγγαρία λέγει ότι θα πρέπει να προστατεύονται κάποια χαρακτηριστικά προϊόντα για ε, ένα λαό και ένα έθνος. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που τόσος πολλοί κόσμος ενδιαφέρεται για την Ουγγαρία αυτό τον καιρό και θεωρούμε σημαντικό να ε, ενδιαφερθούν και για τα ουγγρικά προϊόντα. που είναι πάρα πολύ ε, παραδοσιακά και πάρα πολύ χρήσιμα. να, μην μιλήσω για τον Χούνιαντι τον Πούσκας, τον ε, πολύ γνωστό προπονητή. Ε, ε, έχουμε όχι μόνο σημαντικά προϊόντα αλλά και σημαντικές προσωπικότητες. Κοιτάξτε, ένα λεπτό σας είπαμε. Ο κύριος Σόλτες έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πιστεύω ότι η προστασία γεωγραφικής ένδειξης και η επέκτασή της και σε μη γεωργικά προϊόντα είναι πολύ θετική, γιατί θα δημιουργήσει μεγαλύτερη διαφάνεια και θα βοηθήσει τους καταναλωτές ε, να κάνουν ε, πιο τεκμηριωμένα και έχοντας καλύτερη επίγνωση κατάσταση στις επιλογές τους. Άλλωστε, η επέκταση αυτή της ε, προστασία γεωγραφικής ένδειξη δεν εξασφαλίζει αυτόματα και την ιχνηλασιμότητα. Η ιχνηλασιμότητα θα εξασφαλιστεί με επιπλέον μέτρα. Θα πρέπει επίση να επικεντρωθούμε σε θέματα ασφάλεια ε, των προϊόντων και ελέγχου τη αγορά. Κάτι άλλο που είναι σημαντικό για του πράσινου ε, αφορά το γεγονό ότι η έκθεση δεν περιλαμβάνει αρκετέ πληροφορίε για, για τα δικαιώματα πνευματική ιδιοκτησία αυτών των νέων προϊόντων. Θα πρέπει να γίνουν κάποιε μελέτε επιπτώσεων για να δούμε σε τι βαθμό η προστασία γεωγραφική ένδειξη και επέκτασή τη σε μη γεωργικά προϊόντα θα έχει κόστο και ποιο θα είναι αυτό το κόστο της επέκτασης. Αυτά ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, λέει ο κύριος Πασπίσιλ. Και εγώ τάχθηκα υπέρ της έκθεση, όπως η συντριπτική πλειοψηφία των συναδέλφων, γιατί πιστεύω ακράδαντα ότι σε μια εποχή που σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωσης έχουμε προστασία των γεωργικών προϊόντων ε, με τη γεωγραφική ένδειξη, είναι λογικό να επεκτείνουμε την προστασία αυτή και σε άλλα προϊόντα που δεν είναι αγροτικά. Επίσης, σε κάθε περιοχή υπάρχουν πολλά ντόπια ε, παραδοσιακά προϊόντα. Γιατί να μην και αυτά υπόψη σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και να εξασφαλιστεί η προστασία τους ε, πανευρωπαϊκά για να μην εμπίπτουν σε 28 διαφορετικά και κατακαιρματισμένα συστήματα προστασίας γεωγραφικής ένδειξης. Άλλωστε, η πρόταση αυτή σε καμία περίπτωση δεν στρεβλώνει ή δεν εμποδίζει τον ανταγωνισμό μεταξύ των παραγωγών. Θα ισχύσει ο ελεύθερο ανταγωνισμό, α μην το ξεχνούμε αυτό και να το υπενθυμίσουμε στου επιχειρηματίε. Η κυρία Μάλετιτ, ευχαριστώ. Και εγώ υπερψήφισα την πρόταση για επέκταση τη προστασία γεωγραφική ένδειξη τη Ευρωπαϊκή Ένωση και σε μη γεωργικά προϊόντα, γιατί και τα μη γεωργικά προϊόντα είναι όπως τα γεωργικά είναι φορείς ε, οικονομικής ανάπτυξης και οικονομικής μεγέθυνσης και εδώ έχουμε μια πολύ καινοτόμα προσέγγιση και πρόθεση της παράδοσης. Έτσι θα προωθήσουμε τις ευρωπαϊκές μας αξίες με τις οποίες συμφωνούμε. Επίσης θα δημιουργήσουμε και θέσεις απασχόλησης, θα στηρίξουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τους βιοτέχνες. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, ιδιαίτερα στην Ήπεθρο αλλά και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές της Ένωσης. Ε, στην Κροατία έχουμε μεγάλη προσφορά τέτοιων ε, προϊόντων και μπορούμε να δείξουμε στην Ευρώπη και στον κόσμο ότι έχουμε ιδιαίτερα και πολύ ποιοτικά, όχι μόνο γεωργικά προϊόντα, όπως είναι τα μανταρίνια, το ζαμπον κούλεν, ε, πατάτες από το ηλίτσκοκ και σουκρούτ μπορούμε να δείξουμε ότι έχουμε και μη γεωργικά προϊόντα που είναι άξια προστασίας και καλό, γι' αυτό τάχθηκε υπέρ τη επέκταση τη προστασία. Ο κύριο Κέλλη. Θέλω να σα εξηγήσω για ποιο λόγο υπερψήφισα την έκθεση αυτή. Πρέπει να σας πω ότι χτες το βράδυ πήγα στη συζήτηση και ήταν προφανέ πως η πλειοψηφία των ευρωβουλευτών ήταν υπέρ. Και το είδαμε αυτό και από τον τρόπο με τον οποίο ψήφισαν. 694 υπέρ. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία πως αυτή η προστασία που προσφέρουμε έχει βοηθήσει ε, τα γεωργικά προϊόντα. Και με τον τρόπο αυτό θα έπρεπε να στηρίξουμε και άλλα, μη γεωργικά. Νομίζω λοιπόν ότι με τον τρόπο αυτό θα μπορούσαμε να προωθήσουμε τις πωλήσει, θα δημιουργούσαμε και θα προστατεύαμε θέσεις εργασίας, θα δημιουργούσαμε πλούτο. Όπως είπε και η εισηγήτρια, ελπίζω πως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα καταβάλει κάθε προσπάθεια έτσι ώστε οι προτάσεις να φτάσουν το συντομότερο δυνατόν. Η κυρία Γράτσι. Ευχαριστώ. Συνάδελφοι, μόλις εγκρίναμε μια έκθεση πρωτοβουλίας χάρη στην οποία τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούν να εισαγάγουν και την ε, γεωγραφική έκθεση για μη γεωργικά προϊόντα. Μέχρι τώρα έχουμε ονομασίες προέλευσης για τυριά, για κρέας κτλ. Και τώρα αυτό θέλουμε να επεκταθεί σε άλλα προϊόντα όπως είναι ε, κάποια ε, προϊόντα όπως ότι το μάρμαρο της Καράρα ή κάποια κρίσταλα ή άλλα προϊόντα κεραμικά. Αυτό το Made in έχει σκαλώσει λοιπόν και είναι κρίμα που ε, το μητρό αυτό, ο κατάλογος ε, γεωγραφικών προελεύσεων ε, δεν είναι δωρεάν. Εμείς θα προτιμούσαμε δωρεάν. Μαμίκινς για ένα λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η γεωγραφική ένδειξη και η επέκτασή της σε μη γεωργικά προϊόντα είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και εκ των ουκ άνευ. Θα βοηθήσει να ε, ενημερώνονται καλύτερα οι καταναλωτές και να ε, επιλέγουν με τα λόγου γνώσεως. για να ξέρουν ε, ότι είναι ποιοτικά τα προϊόντα αυτά ε, η ε, παραγωγή επίσης είναι καταναλωτές και ήδη. Και είναι πολύ σημαντικό να προστατεύουμε την παραδοσιακή μας παραγωγή για να διατηρούμε τον πληθυσμό στην Ήπεθρο και τις θέσεις εργασίας. Στη Λετωνία είναι πάρα πολύ ισχυρές αυτές οι τάσεις, ιδιαίτερα στις πιο φτωχές υπαίθριες ε, περιοχές στην Ανατολική Λετωνία. Ευχαριστώ κύριο Σπόλτσακ. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Και εγώ υπερψήφισα την έκθεση γιατί κατά τη γνώμη μου δεν πρέπει να ξεχνούμε τη σημασία που έχει η προστασία αυτών των προϊόντων που δεν είναι μόνο βιοτεχνικά αλλά καλύπτει μια, ένα ευρύτατο φάσμα προϊόντων. Επίσης, δεν θα πρέπει να ξεχνούμε την ενημέρωση και την προστασία του καταναλωτή. Παρέχονται πολύ περισσότερες πληροφορίες στους καταναλωτές για τα τοπικά αυτά προϊόντα. Καλό θα ήταν λοιπόν τέτοια προστασία να έχει πανευρωπαϊκό χαρακτήρα. Γιατί αν ε, δώσουμε την δέουσα αξία στο βιοτεχνικό κλάδο, θα στηρίξουμε ουσιαστικά την παρουσία του και διεθνώς. Γι' αυτό και θα έλεγα ότι καλό θα ήταν να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις για τα TRIPS. Είναι σημαντικό για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο κύριος Μαολού. Ευχαριστώ. Είναι πολύ σημαντική η έκθεση που ψηφίσαμε σήμερα και ελπίζω ότι και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα αναλάβει ε, ταχύτατα δράση προτείνοντας ένα νομοθετικό πλαίσιο για την πρόταση αυτή. Στην Ιταλία έχουμε μακρά παράδοση με τέτοια τοπικά προϊόντα. Χρειαζόμαστε λοιπόν αυτό το σήμα Made in, όχι μόνο τα γεωργικά, αλλά και για άλλα προϊόντα. Θα βοηθήσουμε έτσι τις επιχειρήσεις που έχουν να αντιμετωπίσουν την, τον παγκόσμιο ανταγωνισμό. Γιατί οι τελικές επιχειρήσεις ε, χαρακτηρίζονται για τα πολυποιωτικά προϊόντα τους. Ωραία, περάσαμε, ε, ολοκληρώσαμε τις επεξηγήσεις ψήφου για την έκθεση Ροζιέρ. Περνάμε στην έκθεση Μιχαήλωβα. κυρία Μόρβα, ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ. Είναι προφανές και αυτονόητο ότι υπερψήφισα εγώ ε, να δοθούν περισσότερα κονδύλια από τον κοινοτικό προϋπολογισμό στην Ελλάδα. Αλλά όπως είπα και προηγουμένως, ε, στην τοποθέτησή μου, θέλω να ζητήσω από τους Έλληνες πολίτες να ελέγχονται τα κονδύλια αυτά, πώς δαπανώνται. Και αν βλέπουν ότι ε, χρηματοδοτούνται διεφθαρμένα έργα με κοινοτικά κονδύλια, θα πρέπει αμέσως να το καταγγέλουν. Όπως έπραξα και εγώ προσωπικά όταν διαπίστωσα ότι στην Ουγγαρία υπήρξαν ελάφροχειρίε σε σχέση ε, με ε, κάποιες αγοραπολισίες γεών, διότι διαπίστωσα ότι τα ευρωπαϊκά κονδύλια και ευρωπαϊκές ενισχύσεις είναι αντικείμενο χειραγώγησης και ε, σε ό,τι αφορά τις εκμισθώσεις γεών και το κατήγγυλα. Ε, απευθύνθηκα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το διαβίβασα αρμοδίως και εκείνοι το έδωσαν στην Όλαφ. Η Πρόεδρος, θα σας παρακαλώ να σέβεστε το χρόνο Κυρία Μάλετιτς. Ευχαριστώ. Σήμερα υπερψηφίσαμε συγκεκριμένα ειδικά μέτρα έκτακτη νομοθεσία για να βοηθήσουμε την Ελλάδα να εκταμιεύσει και να απορροφήσει πολύ γρήγορα τα κοινοτικά κονδύλια. μην ξεχνούμε όμω ότι και άλλε χώρε μέλη έχουν προβλήματα με τη χρηματοδότηση των επενδύσεων και των στρατηγικών του σχεδίων και προγραμμάτων και δεν έχουν συχνά τα επαρκή κονδύλια και μέσα για την συγχρηματοδότηση. Γι' αυτό απευθύνω έκκληση προ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, να σκεφτεί πώ θα βοηθήσει τα κράτη-μέλη να εκταμιεύουν πιο γρήγορα τα κοινοτικά κονδύλια και να βοηθήσουμε ιδιαίτερα τα κράτη-μέλη που έχουν μεγάλη στέρηση και για τα οποία υπάρχει και ειδική task force Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Για τις χώρες αυτές που υστερούν θα πρέπει να προστατεύσουμε την όλη νομοθεσία και τους κανόνες ώστε η εφαρμογή των κοινοτικών κονδυλίων να γίνεται πιο γρήγορα και να είναι πιο αποτελεσματική. Επίσης απευθύνουμε έκκληση και στην κυβέρνηση να ε, υιοθετήσει εθνικά μέτρα απλούστευσης γιατί είναι πολλά τα επίπεδα νομοθεσίας που θα πρέπει να διορθωθεί το θέμα αυτό. Ευχαριστώ κύριε Σκέλη ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ. Όταν ήταν εδώ ο κύριο Τσίπρας, μίλησα εκ μέρου του ΕΛΚ και του άσκησα κριτική και του είπα, αν μα παρουσιάσετε ένα σοβαρό πακέτο, εμεί ε, θα συνεργαστούμε μαζί σα. και πρέπει να σα πω το έκανε και έχει ξαναεκλεγεί. Η κατάσταση για την Ελλάδα είναι πολύ δύσκολη. Εμεί, ε, από την Ιρλανδία ξέρουμε πόσο δύσκολο ήταν το πρόγραμμα λιτότητα, αλλά το ακολουθήσαμε και στη χώρα μα βελτιώνεται η κατάσταση. Ελπίζω το ίδιο να συμβεί και στην Ελλάδα. Πρέπει να γίνει κάθε προσπάθεια να βοηθηθούν οι Έλληνε και αν μπορούμε μέσω των διαστατικών επιδοτικών ταμείων να είμαστε λιγότερο αυστηροί με την Ελλάδα, τότε έχουμε την υποχρέωση να το κάνουμε. Αναγνωρίζουμε πως η Ελλάδα αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζει πολύ μεγάλο βάρος με το ε, μεταναστευτικό. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να τους βοηθήσουμε όσο μπορούμε και αυτός είναι ένας πολύ καλός τρόπος, ένα πρώτο βήμα. Ο κύριος Ποσπίλ πρώτος. Ευχαριστώ πολύ. Να σας πω πως ε, εγώ έχω ασχοληθεί με το θέμα και θα ήθελα να στηρίξω την Ελλάδα και κυρίως σε μια κατάσταση την οποία διανύει αυτή τη στιγμή που είναι δύσκολη. Και πιστεύω πως θα πρέπει να θεωρήσουμε πως αυτό είναι μια εξαίρεση που προσφέρουμε στην Ελλάδα, ε, μια εξαίρεση την οποία διατυπώνουμε ε, για το μέλλον μέχρι το 2020 και θα το επαναλάβουμε και τον Ιούνιο. Ε, πρέπει να σας πω πως στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Συνόδου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε υλικό και προτάσεις που έκλεινε την προγραμματική περίοδο 2007-2013 ε, και ξαφνικά καταφτάνει μια αναδρομική πρόταση η οποία ενδεχομένως να περιπλέξει τα πράγματα. Νομίζω πως αν θέλουμε να ψηφίσουμε ε, για βοήθεια να είναι βοήθεια για το μέλλον έτσι ώστε να μην το κάνουμε μετά την περάτωση του προγράμματος. Ο κύριος Μάμενκιν είναι ο επόμενος ομιλητής. Ευχαριστώ. Η πρόταση αυτή αφορά στην έγκριση ειδικών μέτρων προς την Ελλάδα προκειμένου να αυξηθεί η δυνατότητα απορρόφησης. Έχουμε ουσιαστικά χρηματοδότηση 100% από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης ε, έχουμε και ε, μια επιπλέον βοήθεια για την περίοδο 2014-2020, κυρίως σε επενδυτικά προγράμματα. Η προσφορά βοήθειας ε, είναι απαραίτητη για να αυξηθεί και η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας. Βέβαια, βασικός στόχος είναι η συνδρομή μας προς την ελληνική κυβέρνηση για να εφαρμόσει τις μεταρρυθμίσεις και να μπορέσει η Ελλάδα να επιστρέψει στο δρόμο και στην κατηγορία των πιο προοδευτικών και ανεπτυγμένων χωρών του κόσμου. Είμαι υπέρ, ε, τάχθηκα υπέρ αυτής της ε, έκθεσης. Ο κύριος Πόλτσακ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ υπερψήφισα την έκθεση που ζητά την παροχή συγκεκριμένης βοήθειας προς την Ελλάδα. Ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Τσίπρας, Είχε αναφερθεί και στα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η χώρα αυτή και νομίζω ότι η συγκεκριμένη έκθεση αποτελεί σημαντική χειρονομία ευρωπαϊκής αλληλεγγύης. Και τα 5 εκατομμύρια ευρώ που θα ληφθούν από τα αποθεματικά για να ληφθεί υπόψη ο φετινός αντίκτυπος και ο αντίκτυπος που θα έχει του χρόνου το προσφυγικό θέμα και δεδομένη της ε, οικονομικής κατάστασης και του νομοθετικού πλαισίου κρίθηκε αναγκαίο να θεσπιστούν αυτά τα ειδικά μέτρα. Εγώ θα προτιμούσα να είχαμε συνδέσει την παροχή των κονδυλίων αυτών με την ε, εφαρμογή ορισμένων έκθεση διότι τα ληφθούν για την στήριξη της Ελλάδας είναι αποφασιστικά μια χώρα η οποία υπέφερε και υποφέρει ακριβώς λόγω των μνημονίων. τα μνημόνια φτωχοποίησαν την ελλάδα. ταυτόχρονα τα μνημόνια επέβαλαν την μείωση των δημοσίων επενδύσεων. επομένως χωρίς δημόσιες επενδύσεις δεν μπορούσε να υπάρξει συγχρηματοδότηση από πλευράς ελλάδας άρα δεν μπορούσε να γίνει και η απορρόφηση των κοινοτικών κονδυλίων. ξεκάθαρα λοιπόν τα μέτρα αυτά ήταν αποφασιστικά προκειμένου να προχωρήσουμε. να προχωρήσουμε σε μια φάση που η ίδια η ευρωπαϊκή ένωση μέσω της τρόικας έχει φτωχοποιήσει την ελλάδα. γι' αυτό λέμε και την παροιμία να σε κάψω γιάννη να σ' αλείψω μέλι δηλαδή έρχεται τώρα η ευρωπαϊκή ένωση να συμπληρώσει να βοηθήσει τον ελληνικό λαό έστω και περιορισμένα για να ανακουφιστεί από αυτές τις επιθετικές και άδικες πολιτικές του ίδιου του μνημονίου. ευχαριστώ. Πάμε τώρα στην έκθεση Θεοχάρους και σε επεξηγής ψήφου και θα δώσω το λόγο στον κύριο Πόσπισελ για ένα λεπτό. Ναι. Ε, ε, ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Εγώ υποστήριξα την έκθεση αυτή και την υπερψήφισα. Είμαι από την Τσεχική Δημοκρατία και ξέρετε ότι εμείς υποστηρίζουμε τις αναπτυσσόμενες χώρες με τρόπο ενεργό και είμαστε πολύ δραστήριοι. Ήδη από το 2013 και μέχρι το 2020 έχει διπλασιαστεί ε, η χρηματοδότησή μας στην αναπτυξιακή βοήθεια από την Τσεχική Δημοκρατία. Και αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να πιάνει τόπο αυτή η βοήθεια, να χρησιμοποιείται σωστά για ουσιαστική συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση και να μην πέφτει στα χέρια των κυβερνήσεων και τελικά στις τσέπες τους. Γιατί πολλές φορές είναι αμφιλεγόμενη η ε, κατάληξη της βοήθειας αυτής που δεν φτάνει στους τελικούς δικαιούχους. Η φιλοσοφία λοιπόν της έκθεσης είναι σωστή, γι' αυτό και την υποστήριξα. Ο κύριος Κέλλη, ευχαριστώ και πάλι πρόεδρε. Υπερψήφισα και εγώ την έκθεση ε, και με χαρά. Όπως και τα περισσότερα ε, μέλη του Κοινοβουλίου, 506 ε, ψήφους ε, πήρε η έκθεση κυρία Θεοχάρος. Γιατί σε τοπικό επίπεδο γίνεται αυτή η δουλειά. Οι αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης είναι πιο κοντά στον πολίτη και βελτιώνουν τη ζωή τους. Και ο κόσμος το αναγνωρίζει αυτό και ταυτίζεται και με την αυτοδιοίκηση. Ε, είναι μακριά οι κεντρικές κυβερνήσεις, πολλές φορές δικτάτορες και τα χρήματα που τους προσφέρουμε ε, πηγαίνουν σε λάθος κατεύθυνση και σε λάθος χέρια. Είναι καλή η έκθεση αυτή και θα βοηθήσει τις αναπτυσσόμενες χώρες να χρησιμοποιήσουν με το σωστό τρόπο τα κονδύλια αυτά. Ο κύριος Μαμέκινς. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Όπως όλοι γνωρίζουμε η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο υπαριθμόν ένα δωρητή αναπτυξιακή βοήθεια στον κόσμο, καθώ είναι και από τι πλουσιότερε περιφέρειε του κόσμου. Είναι καθήκον μα λοιπόν να βοηθούμε τι στοχότερε περιφέρειες. Ένα τρόπο για να γίνει αυτό είναι με την αναπτυξιακή βοήθεια, αλλά μέσω των ε, οργανισμών τοπική αυτοδιοίκηση. Ε, ε, ε, στην περιφέρεια κρίνονται αυτά τα ζητήματα, μακριά από τις πρωτεύουσε. Εκεί γίνεται η περισσότερη ανάπτυξη σε οποιαδήποτε χώρα. Γι' αυτό θα πρέπει και εμείς να μοιραζόμαστε τον πλούτο μας με τις φτωχές ε, χώρες και περιφέρειες. Αυτό ισχύει για όλες τις χώρες, όχι μόνο για τις αναπτυσσόμενες, αλλά και η δική μου χώρα, η Λετωνία, ε, ε, ε, βλέπει τεράστιες διαφορές ανάμεσα στην πρωτεύουσα Ρήγα και την περιφέρεια Φλάτκαλα που είναι η πιο φτωχή. Ευχαριστώ πολύ ο κύριος Πόλτσακ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Υποστήριξα και εγώ την έκθεση της κυρίας Θεοχάρους που είναι και από την πολιτική μας ομάδα. Όχι επειδή θεωρώ μόνο ότι είναι σημαντική δουλειά της τοπικής αυτοδιοίκησης. Εκτός αυτού ε, θεωρώ ότι πιάνει και τόπο ε, από πολιτικής πλευράς και όταν καλούμε να υλοποιήσουμε τους πολιτικούς στόχους της Ένωσης και προστατεύει η τοπική αυτοδιοίκηση τις αξίες και τις αρχές μας πολύ περισσότερο από τις κεντρικές κυβερνήσεις. Αφήστε δε και την αρχή της επικουρικότητας ή της αναλογικότητας ε, που εφαρμόζει τοπική. Αυτό πραγματικά αξίζει την υποστήριξη και την προσοχή μας. Επιπλέον θα ήθελα να σας πω ότι είναι απολύτως σημαντικό να αναγνωρίσουμε το ρόλο της τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά να είναι και στο ύψος ε, των υποχρεώσεων και των καθηκόντων της. Δούμε λοιπόν το πώς ε, χρέο έχουν οι κυβερνήσεις ε, η τοπική αυτοδιοίκηση έχει μικρή συμμετοχή. Στην Τσεχική Δημοκρατία είναι μόλις το 10% ε, η συμμετοχή της τοπικής αυτοδιοίκησης στο χρέος. Και αυτό έχει τη σημασία του ε, για το πώς διαχειρίζονται πολύ χειρότερα οι κεντρικές κυβερνήσεις από τις τοπικές. Η κυρία Μόρβα, ευχαριστώ πολύ πρόεδρε. Και πάλι πρέπει να σας πω ότι υπερψήφισα την έκθεση για τους ίδιους ακριβώς λόγους με την περασμένη φορά. Πρόκειται για ευρωπαϊκά κονδύλια που θα πρέπει να την χάνουν της διαχείρισης και ε, δεν θα πρέπει να βασιλεύει εκεί ο νεποτισμός και οι κρυφές συναλλαγές. Και θέλω να επανέλθω εκεί που σταμάτησα ε, στην προηγούμενη έκθεση, διότι αυτό ακριβώς συνέβη στην Ουγγαρία. Με αυτές τις γεωργικές ενισχύσεις που σας έλεγα και τις ατασταλίες θα ήθελα λοιπόν να καλέσω όλους και στην Ευρώπη και στην Αφρική να προσέχουν πώς ε, ποιος διαχειρίζεται αυτά τα κονδύλια και όταν υπάρχουν αποδείξεις για αλαφροχειρίες και αταστηλίες να απευθύνονται στις αρμόδιες αρχές. Εμείς απευθυνθήκαμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Επιτροπή το διαβίβασε στην Όλαφ, η οποία Όλαφ έχει επιληφθεί του θέματος και ε, μπορούμε να καταλάβουμε τι γίνεται. Τελειώνει εδώ η επεξήγηση ψήφων τη συνεδρίαση μέχρι τις 3 το μεσημέρι. Ευχαριστώ.